και να ενισχύσουμε τις προσπάθειες μεταρρύθμιση που κάνει η Σερβία, ώστε η χώρα αυτή να μπορέσει όσο γίνεται πιο γρήγορα να περάσει τις διαπραγματεύσει μαζί μας. Έχουμε το σχέδιο αυτοψηφίσματο με το οποίο κλείνει η συζήτηση. Αύριο θα γίνει ψηφοφορία στις 11.30. Τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση για την διεύρυνση σε ό,τι αφορά το Κωσυφοπέδιο. Έχουμε δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή. Και πάλι εκ μέρου του Συμβουλίου το λόγο έχει ο Υπουργό, ο κύριο Νικολάη Βάνεν. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, κύριε Επίτροπε. Σε ό,τι αφορά το κοσυφοπαίδιο θα πρέπει να πω με σαφήνεια ότι είμαι αισιόδοξο για την κατάσταση όπως ε, εξελίχθηκε μετά από την υποβολή της έκθεσης ε, προόδου του 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Συμβούλιο και τα συμπεράσματα 28 Φεβρουαρίου φέτος αποτυπώνουν τις σημαντικές ε, προσπάθειες που έγιναν και από τη Σερβία αλλά και από το 25 στο διάλογο τον οποίο διευκολύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω ξέρετε, το Συμβούλιο τον προηγούμενο Δεκέμβριο καλωσόρισε τη δέσμευση του 25 στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα συμπεριλαμβανομένων ε, των ε, διαρκών προσπαθειών σε τομείς όπως οι θεωρήσεις, το εμπόριο και το δικαστικό σύστημα, καθώς και σε ό,τι αφορά την ίδρυση ενός Εθνικού Συμβουλίου για την ε, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλωσόρισε την καλύτερη ενσωμάτωση των Σέρβων νότια του ποταμού Ήμπαρ. Παράλληλα, το Συμβούλιο σημειώνει την περιορισμένη πρόοδο που σημειώθηκε σε ό,τι αφορά τη μεταρρυθμιστική ατζέντα σε ένα έτος το οποίο σημειώθηκε από την διεξαγωγή εκλογών και το Κοινοβούλιο ε, ζήτησε από το 25 να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την ε, ε, διαδικασία διεξαγωγή των εκλογών. Το Κωσυφοπέδιο επίσης ενθαρρύνθηκε να βελτιώσει την κατάσταση σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, σε στενή συνεργασία με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Το Συμβούλιο σημειώνει την ανάγκη για μεγάλε προσπάθειε από πλευρά των αρχών σε ό,τι αφορά την ενίσχυση τη δημόσια διοίκηση και τη μεταρρύθμιση και τη ενίσχυση του κράτου δικαίου. Χρειάζεται χρειάστηκαν στοιχεία για να καταδείξουν ότι το οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά αντιμετωπίζουν και ότι γίνεται πρόοδο σε ό,τι αφορά την δικαστική μεταρρύθμιση και την προστασία τη ελευθερία τη έκφραση. Το Συμβούλιο επίση κάλεσε το Κωσυφοπαίδιο να ξεκινήσει την ατζέντα για το Βόρειο Κωσυφοπαίδιο. Πέρα από αυτέ τι απαιτήσει, το Συμβούλιο τόνισε τη βασική σημασία του διαλόγου Βαλιγραδίου και Πρίστινα σαν ένα, μια διαδικασία εξίσου μεγάλη σημασία και για τη Σερβία και για το Κωσυφοπέδιο. Επίση, το Συμβούλιο κάλεσε και τι δύο πλευρέ να συνεχίσουν ε, επικοδομητικά να συνεργάζονται σε πολλού τομεί, από την ελευθερία και μετακίνηση των ατόμων, μέσα στην τελωνία, από τα κτηματολόγια μέχρι την εφαρμογή τη ε, κοινή διαχείριση των σημείων διασταύρωση. Αυτή η έκκληση ακούστηκε και από το Βελιγράδι και από την Πρίστινα. Έγινε, έγιναν σημαντικές πρόοδοι τους τελευταίους μήνες και αυτό έδωσε πολιτικό, αν θέλετε, κουράγιο και στις δύο πρωτεύουσε. Ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη που καταδεικνύει τη σημασία και τη δύναμη της διαδικασίας ε, ε, διαβρυνσής για την πρόθεση των μεταρρυθμίσεων. Επίσης και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχε ανταπόκριση στις προσπάθειες αυτές. Ο διάλογος για τις θεωρήσεις ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012 και επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ξεκινήσει διάλογο για το κράτος δικαίου, καθώς και μία μελέτη εφικτότητας για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κωσυφοπεδίου. Αυτά είναι σημαντικές, ε, σημαντικά βήματα, Πρόεδρε, αξιόλυμοι βουλευτές, Επίτροπε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το μέλλον του Κωσυφοπεδίου είναι στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλή εφαρμογή των ε, συμφωνιών μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα θα οδηγήσει τη Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο πέρα-πέρα στο μονοπάτι τους, αν θέλετε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφετέρου, πολλές είναι οι προκλήσεις που παραμένουν για την ηγεσία στο Κωσυφοπαίδιο, μεταξύ άλλων και στον εγχώριο τομέα. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να ε, βοηθήσει και ελπίζω να αφιερωθούν πιο πολλοί πόροι για να υποστηριχθούν οι πρωτοβουλίες από τις Βρυξέλλες καθώς και ε, του νέου ειδικού εντεταλμένου που ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις πριν από κάποιες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ, Υπουργέ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον ε, Επίτροπο Φίλα, εξ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε αξιότιμοι ευρωβουλευτές κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να έρθω να συζητήσουμε εδώ για το Κωσυφοπαίδιο. Σα είμαι ευγνώμων επίσης για την στήριξή σας στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το Κωσυφοπαίδιο, όπως αυτή φαίνεται και στην έκθεση που συζητάμε σήμερα. Είμαι ευγνώμων επίσης και στην εισηγήτριά σας την κυρία Λούνα Τσεκ για την έκθεση αυτή που είναι καλά ισορροπημένη. Μόλις επέστρεψα από το κοσυφοπέδιο, την Τρίτη, με ιδιαίτερη χαρά βρέθηκα στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου του κοσυφοπεδίου για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργήθηκε το Συμβούλιο αυτό από τον Πρόεδρο Γιατζάκα προκειμένου να αποτελέσει μια βάση για συζήτηση και προκειμένου το κοσυφοπέδιο να μπει στο δρόμο της Ευρώπης. Στην ομιλία μου εκεί υπογράμμισα ότι είναι πολύ βασικό στο Συμβούλιο να συμμετέχουν όλες οι πλευρές του πολιτικού φάσματος του κοσυφοπεδίου και να στηρίζεται από όλες τις πλευρές. Το Συμβούλιο πρέπει να πετύχει ευρεία συνένεση και να φροντίσει για την συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας. Μόνο με τη στήριξη και τη δέσμευση όλων των πολιτικών δυνάμεων και κοινοτήτων θα μπορέσει το κοσυφοπέδιο να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται και ο δρόμος του για την Ευρώπη να καταλήξει θετικά. Απαιτείται η στήριξη και η δέσμευση της κοινωνίας του κοσυφοπεδίου ολόκληρης, γιατί από τη φύση της η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να αφήνει κανέναν απ' έξω. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βάλουμε πιο κοντά το κοσυφοπαίδιο στο δρόμο αυτό για ένταξη. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τη 28 η Φεβρουαρίου επιβεβαίωσε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ξεκινήσει μια μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την Συμφωνία Σταθερότητας και σύνδεση με το Κωσυφοπαίδιο. Αυτό αποτελεί ένα νέο ξεκίνημα όσον αφορά τι σχέσει τη Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κωσυφοπαίδιο. Η έγκριση επίσης του Συμβουλίου φέρνει πιο κοντά το κοσυφοπέδιο στην ε, πολιτική πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά ε, Βαλκάνια. Στόχος της μελέτης κοπιμότητας ε, πάντως είναι να κάνει μία πλήρη και σε βάθος ανάλυση όσον αφορά το κατά πόσο είναι το κοσυφοπαίδιο έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και να θέσει σε εφαρμογή τελικά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Σύνδεσης, το οποίο αποτελεί και τη νομική βάση για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και ένα σταθμό στην πορεία προς την ένταξη. Η μελέτη θα επικεντρωθεί στις πολιτικές, οικονομικές και νομικές επιτυχίες όσον αφορά το κατά πόσο το κοσμοπέδιο είναι έτοιμο για την συμφωνία αυτή σταθερότητα και σύνδεσης. Η επίσκεψή μου στο κοσυφοπέδιο ακριβώς κατέδειξε και την αρχή του έργου αυτού. Η μελέτη σκοπιμότητας επιπλέον αποτελεί ένα στοιχείο κλειδί όσον ε, αφορά την ε, ήδη φιλόδοξη ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κωσυφοπαίδιο. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία τώρα. Πρώτα απ' όλα ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε το χάρτη πορείας για την ελευθέρωση ε, των θεωρήσεων. Δεύτερον, ότι θα μπορέσουμε πολύ γρήγορα να υποβάλουμε πρόταση για μια συμφωνία πλαίσιο που θα επιδεύει στο Κωσυφοπέδιο να συμμετέχει στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτο, στις 30 Μαϊού θα ξεκινήσω έναν διαρθρωτικό διάλογο όσον αφορά το κράτος δικαίου. Τέταρτον, θα στηρίξουμε την αίτηση του Κωσυφοπαιδίου προκειμένου να γίνει μέλο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Νοικοδόμηση και ανάπτυξη εφόσον το Κωσυφοπέδιο υποβάλλει την αίτηση αυτή. Πέμπτο, είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε μία συμμετοχική και μακρά ε, ατζέντα όσον αφορά το Βόρειο Κόσοβο. Επιτρέψτε μου τώρα να επιβεβαιώσω την δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ Κωσυφοποδίου. Τελευταίε εβδομάδε έδειξαν ότι δεν πρόκειται για κενά λόγια μόνο, αλλά ότι στηρίζονται και από συγκεκριμένε δράσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί υπέρ του κοσυφοπεδίου. 2012 είναι η χρονιά που πρέπει να αποτελέσει τη χρονιά των ευκαιριών και πιστεύω ότι μπορώ να βασιστώ στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε η ευκαιρία αυτή να γίνει και πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Επίτροπε, τώρα εκ μέρους των πολιτικών ομάδων θα ακούσουμε τους διάφορους ομιλητές. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την κυρία Ελρίκε Λούνατσεκ εκ μέρους των Πρασίνων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και εσάς ε, κύριε Φούλε και τον κύριο Βάνεν εκ μέρους της Προεδρίας. Εφέτος η έκθεσή μου έχει ως ε, στόχο να στείλω ένα χειρό μήνυμα στους πολίτες ε, του Κωσοπεδίου ότι το μέλλον τους είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση αναγνωρίζει τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους τελευταίους, τον τελευταίο μήνα και χρόνο ε, μιλήσαμε για τον οδικό χάρτη, για την κατάργηση της ε, θεώρησης. Ο οδικός χάρτης θα υπάρξει αυτή την άνοιξη. Ο διάλογος ανάμεσα στην Πριστίνα και το Βελιγράδι, ανάμεσα στο Κοσοπέδιο και τη Σερβία, οδήγησε σε κάποια θετικά αποτελέσματα και πρέπει να συνεχιστεί μετά τις εκλογές ε, στη Σερβία. Αποτέλεσμα, περιφερειακή συνεργασία. Τώρα το Κοσμοπέδιο μπορεί να συμμετέχει αυτόνομα σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και η Συμφωνία για τη Διαχείριση των Συνόρων. Για πρώτη φορά έχουμε διμερή συμφωνία ανάμεσα στα δύο κράτη. Βέβαια, καλό τη Σερβία να υπογράψει τη συμφωνία αυτή όπως υποσχέθηκε. Και επίση, ε, κύριε Φίλε, εχθέ ε, με την επίσκεψή σα ε, δρομολογήσατε τη μελέτη σκοπιμότητα. Είναι το πρώτο βήμα για την περαιτέρω σταθεροποίηση του κοσφοπεδίου. Εγώ αναφέρομαι στα, στις πέντε οντότητες, ε, μάλλον στα πέντε κράτη που πρέπει να αναγνωρίσουν το κοσμοπέδιο, γιατί με τον τρόπο αυτό οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περισσότερο αποτελεσματικές. Βέβαια υπάρχουν ακόμα προκλήσεις στο ίδιο το κοσμοπέδιο, αγώνας κατά του οργανωμένου εγκλήματος, η ε, δημιουργία κοινωνικής οικονομίας, κοινωνική ανάπτυξη, ώστε οι άνθρωποι να θέλουν να δουλέψουν στη χώρα τους. Ε, μεταρρύθμιση εκλογική έτσι ώστε ε, να βρεθούν στην, ε, στα δικαστήρια, στη δικαιοσύνη, ενώπιον της δικαιοσύνης, ως παραβίασαν τον εκλογικό νόμο κατά τις ε, τελευταίες εκλογές. Επίσης, η Πριστίνα πρέπει να απευθυνθεί στους Σέρβους του Βορρά, να έχει τοπική αυτοδιοίκηση σε μεγάλο βαθμό αυτονομία. Καλείται επίσης η Σερβία από το να οργανώσει τοπικέ εκλογές στον Βορρά. Αυτό είναι κατά του διεθνού ε, δικαίου και δεν συμβαδίζει με το ψήφισμα 1244. Να μην έχει επίσης παράλληλε δομέ η Σερβία. Ελπίζω η έκθεσή μου να τύχει ευρεία υποστήριξης ε, και με τις ε, τροπολογίες που κατατέθηκαν, γιατί η πρώτη μου έκθεση ήταν πριν από δύο μήνες και έκτοτε συνέβησαν πάρα πολλά. Εκ μέρου ε, λοιπόν του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, ο κύριο Πόσελτ. Ε, Φέτο έχουν περάσει 100 χρόνια από τον πρώτο πόλεμο στα Βαλκάνια. Ε, αυτά που συνέβησαν τότε είναι τεκμηριωμένα σε στοιχεία του Λοφχόντλιχ, Φρόντλιχ, του Σοσιαλδημοκράτη και πολλών άλλων. Είχαμε 86 χρόνια καταπίεσης και τέλος την προσπάθεια γενοκτονίας από το Μιλόσεβιτς. Εδώ και 12 χρόνια οι Κωσοβάροι έχουν πλέον την ευκαιρία να συστήσουν ευρωπαϊκό δημοκρατικό κράτος. Βέβαια έχουν πολλά προβλήματα, αλλά έχουν προσφέρει, έχουν επιτύχει πάρα πολλά. Σήμερα καλούμεθα να το αναγνωρίσουμε αυτό και να του στηρίξουμε στον δρόμο του στο μέλλον. Ε, ξεκάθαρα λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ της ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό την Κυριακή επισκέφτηκα για τη Σερβία. Όμως θέλω δικαιοσύνη και για το Κοσμοπέδιο. Η Σερβία πήρε την ιδιότητα του υποψηφίου κράτους. Ε, ε, το Κοσμοπέδιο δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί από πέντε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ε, στο Κοσμοπέδιο έχουμε περιορισμένες εκθέσεις και έδρες με περιορισμένες αρμοδιότητες λόγω του σχεδίου Αχτισάρη. Μετά τις τελευταίες εκλογές υπάρχει κίνδυνος οι Αλβανοί να μην έχουν ούτε έναν εκπρόσωπο στο Κοινοβούλιο. Οι Σέρβοι έχουν στο Κοσμοπέδιο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να επικρατήσει η σύνεση και οι δύο πλευρές να αντιμετωπίζουν τις ίδιες προϋποθέσεις ε, στον δρόμο τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν νέες συμφωνίες ανάμεσα ε, εννέα μάλλον συμφωνήσαν ανάμεσα στην Πρίστινα και το ε, Οι μισές έχουν υπογραφεί και δεν εφαρμόζονται. Θέλουμε λοιπόν και πράξεις, όχι μόνο λόγια. Θέλουμε πράξεις πριν από τις εκλογές στη Σερβία και όχι μετά ε, εκ των υστέρων να διαψευθούν οι ελπίδες μας. Δεν θέλουμε το διαμελισμό του Κοσμοπαιδίου. Δεν θέλουμε να ξαναξεκινήσει το θέμα της οντότητάς του. Θέλουμε να έχουμε μια νεόκοπη ε, ευρωπαϊκή δημοκρατία. Επόμενη ομάδα, σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Παντσέρη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κυρία Λούνατσεκ πραγματικά έκανε πολύ καλή δουλειά και πιστεύω ότι η σταθεροποίηση της δημοκρατίας στο Κωσοπαίδιο είναι ένας πολύ σημαντικός παράγων. Ο δικός μας στόχος είναι να ενθαρρύνουμε τις αρχές στην Πρίστινα και ποκινούμε τις πολιτικές δυνάμεις ε, να ακολουθήσουμε τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις που είναι σε θέση να εξυγχρονίσουν τη χώρα και να ανοίξουν μια νέα φάση στην ε, πολιτική και κοινωνική ζωή του Κωσυφοπεδίου. Υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα προς επίλυση. Τα υπενθύμησε το Συμβούλιο προηγουμένως και πρέπει να αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα. Κυρίως ε, πρέπει να αντιμετωπιστούν με την απαραίτητη συνέπεια εκ μέρου των αρχών του κοσφοπεδίου. Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση εξελίσσεται. Ε, χαιρετίζουμε λοιπόν ε, την ιστορική συμφωνία ανάμεσα στο Βελιγράδι και την Πρίστινα όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία και την εκπροσώπηση του κοσοπεδίου στα περιφερειακά φόρουμ. Όλα αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων και είναι ένα σημαντικό στοιχείο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Επίτροπος κ. Φίλου είπε ότι είναι θετικό το ότι η Κομισιόν ξεκίνησε μελέτη σκοπιμότητας που να έχει σχέση τη δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοσοπεδίου. Πρέπει συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, γιατί ο δρόμος αυτός δεν είναι μόνο για τη Σερβία και το Κοσμοπέδιο, όχι μόνο διότι μπορούν να έρθουν πιο κοντά αυτές οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά διότι κυρίως θα βοηθήσει όλο αυτό να ξεπεραστεί η δυσπιστία απέναντι στο Κοσμοπέδιο εκ μέρους εκείνων των κρατών που δεν το έχουν καν αναγνωρίσει. Υπάρχει λοιπόν δουλειά από την Ευρώπη, αλλά υπάρχει και δουλειά στο επίπεδο των Κοσοβάρων για να μπορέσουν να επιτύχουν αυτούς τους ε, στόχους τους. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ε, φιλελεύθερη, ο κύριος Κάτσιν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, ευχαριστώ πολύ την κυρία Λούνερτσεκ για μια τόσο καλά ισορροπημένη έκθεση. Οι κάτοικοι του Κωσοφοπεδίου πήραν κάποια καλά νέα επιτέλους από τις Βρυξέλλες. Η μελέτη σκοπιμότητας ξεκινάει, όπως επίσης και οι εργασίες για τις θεωρήσεις. Πρέπει να καθησυχάσουμε τους κατοίκους του Κωσοφοπεδίου γι' αυτό και να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να σταματήσει αυτό το εμπόδιο που έχει να κάνει με τις θεωρήσεις και τα ταξίδια των κατοίκων του Κωσοφοπεδίου στην περιοχή Σέγγεν. Έχει ξεκινήσει το ο επικοδομητικό διάλογο με την Σερβία. Καλή την πίστη και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ο διάλογο ανάμεσα στο Βελιγράδι είναι προς, ε, με το Βελιγράδι είναι προ το συμφέρον του Κωσυφοπεδίου, του πολίτε του και την οικονομία του. Και οι δύο πλευρέ όμω πρέπει να μπουν στο διάλογο αυτό. Το Κωσυφοπέδιο χρειάζεται οπωσδήποτε διάλογο ανάμεσα στην σερβική κοινότητα στο βορρά του Κωσυφοπεδίου και τους Σέρβους που ζουν στο νότιο τμήμα του ποταμού Ιμπάρ ο πολιτισμός ο σερβικός είναι έντονα παρόν στο κοσυφοπέδιο και δεν πρέπει να υπάρχουν εκεί χάσματα. Η Πριστίνα τώρα πρέπει να στραφεί προς τη σερβική κοινότητα στον Βορρά και να ενθαρρύνει την ένταξή του στο ευρύτερο κοσυφοπέδιο. Το Βελιγράδι πρέπει να σταματήσει πια να μιλάει για έναν Βορρά στον οποίο κυριαρχεί η Σερβία διότι ότι κάποτε το μέρος αυτό de facto θα αποτελέσει και πάλι κομμάτι της Σερβίας. Αυτό δεν είναι δυνατόν και πρέπει οι χώρες μέλη να βοηθήσουν να αποκατασταθεί και η κατάσταση. Αυτό όμω που έχει περισσότερο σημασία για το μέλλον του Κωσυφοπεδίου είναι η Πριστίνα να ξεκινήσει διάλογο με τον εαυτό της η συστημική διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα αποτελούν μάστιγα στην οικονομία του κοσφοπεδίου και στο κράτο δικαίου. Πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα για να καταπολεμηθεί το έγκλημα. Συγκεκριμένα αποτελέσματα λοιπόν θέλουμε ώστε το κοσφοπεδίο να πετύχει τη Συμφωνία Σταθερότητα και Σύνδεση γρήγορα. Η πολιτική βούληση είναι πολύ σημαντική για να το πετύχουν. Ευχαριστούμε. Και τώρα από την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά για ένα λεπτό ο κύριος Αγκουράκης, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Το ψήφισμα προωθεί την υπεριαλιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιδιώξεις των μονοπωλίων στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι μια περίοδος βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης και οξύτατων υπεριαλιστικών ανταγωνισμών για αγορές και σφαίρες επιρροής. Το ψήφισμα στηρίζει την επιβολή των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, την καταλήστευση του φυσικού πλούτου του Κωσόβου, την όξυνση της ανεργίας και της φτώχειας. Εγκαλεί προκλητικά τους κατοίκους του Βορείου Κωσόβου που αντιστέκονται στι κατοχικέ δυνάμει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την διαιώνιση τη παρουσία των δυνάμεων τη k τη Ulex και τη μεγαλύτερη Αμερικάνικη βάση εκτό ΗΠΑ. Προσπαθεί να επιβάλλει την αναγνώριση ενό προτεκτοράτου του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι δημιούργημα του βρώμικου πολέμου ενάντια στο Ιουγκοσλάβικο λαό, εκβιάζει απροκάλυπτα το σερβικό λαό να αποδεχτεί το διαμελισμό τη χώρα για να αρχίσουν οι διαδικασίε ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει έτσι τους ασκούς του, ασκού του αιώλου για την όξυνση εθνοτικών αντιθέσεων, την υποδάβληση αποσχιστικών κινημάτων και την επαναχάραξη των συνόρων. Δημιουργούνται κίνδυνοι για νικευμένη πολεμική ανάφληξη. Τασόμαστε ενάντια στην παρουσία των ξένων στρατευμάτων στα Βαλκάνια, τασόμαστε για μια Ευρώπη τη ειρήνη και τη φιλία των λαών που δεν μπορεί να είναι ε, παρά μόνο πάνω στα ερήπια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. E Το Κοσμοπέδιο είναι μια χώρα με μεγάλα δομικά προβλήματα που αποδεικνύονται ε, στη σχέση ε, έχουμε ένα σύστημα δικαστικό το οποίο δεν καλύπτει τις ανάγκες ενός δημοκρατικού κράτους. Έχουμε μια δημόσια διοίκηση που είναι σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική. Ε, δεν έχουμε μέσα ενημέρωση, ε, δεν είναι ικανοποιητική προστασία των ε, μειονοτήτων και υπάρχει και σύγκρουση με τις θρησκευτικές παραδόσεις. Η οικονομία είναι πάρα πολύ αδύναμη. Σε όλα αυτά προστίθεται μια εγκληματικότητα που αφορά στο εμπόριο όπλων, κίνηση ατόμων και ναρκωτικών ε, και αυτό αποδεικνύεται και από μέσα ενημέρωσης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2010 καταδίκασε την ε, συμμετοχή του Πρωθυπουργού ε, στο παράνομο εμπόριο οργάνων του σώματος ε, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και βέβαια πρέπει να παρακολουθήσουμε το Κοσμοπέδιο σε αυτό τον δρόμο που έχει χαράξει τον κοινωνικό και τον δημοκρατικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα από τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριε Πόσελτ, ο κύριος Πόσελτ έχει ερώτηση για τον κύριο Προβέρα. Δέχεστε το ερώτημα. Μπλε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Προβέρα αν γνωρίζει ότι στις... Ε, δεν υπάρχει καμία απόδειξη για το εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων. Φυσικά θα πρέπει να υπάρξει έρευνα στο θέμα αυτό, αλλά δεν υπάρχει κανένα αποδεκτικό στοιχείο. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Προβέρα αν το γνωρίζει αυτό ότι δεν υπάρχει αποδεκτικό στοιχείο. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Μισό λεπτό έχετε για την απάντηση, κύριε Προβέρα. Κοιτάξτε, εγώ ξέρω ότι η αιτίαση αυτή του Συμβουλίου τη Ευρώπη αναφέρεται πάρα πολλές ε, φορές στην έκθεση Συμβουλίου της ε, Ευρώπης και αυτή η ειδησία αναφέρθηκε και από τον BBC. Εγώ δεν είμαι δικαστής και δεν ε, εναπόκειται σε μένα να επαληθεύσω δικαστικά ή αλλο πώς το αν ισχύει ή όχι. Όμως η αιτίαση αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι πάρα πολύ βαριά. Προέρχεται από ένα παγκίνως αναγνωρισμένο οργανισμό και νομίζω ότι αξίζει να τον έχουμε κατά έχουμε κατά νου την αιτίαση αυτή. Ευχαριστώ και τώρα θα ακούσουμε του υπόλοιπου ομιλητέ, λέει ο Πρόεδρο, ο κ. Λίζεκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που μπορώ να πω και να αποκαλέσω κύριο Πρόεδρο τον παλιό φίλο μου και επίτροπο, τον Επίτροπο. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση του συγητή είναι μια καλά ισορροπημένη έκθεση, την, η οποία αξίζει της υποστήριξής μας και καταδεικνύει την μεγάλη δέσμευση και την εις βάθος γνώση του εισηγητή για όσα συμβαίνουν στο κοσυφοπαίδιο, γιατί ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο θέμα το κοσυφοπαίδιο. Αποτελεί ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα, το οποίο θα αποτελέσει και μία μεγάλη πρόκληση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για όλη την ε, διεθνή κοινότητα, γιατί δεν είμαστε οι μόνοι που ενδιαφερόμαστε για την μεταρρύθμιση της χώρας αυτής. Θα ήθελα να πω ότι καλωσορίζω την έκθεση που αναφέρει ότι το κοσυφοπαίδιο έχει πετύχει πολλά σε ό,τι αφορά την ε, αναδιοργάνωση του πολιτικού και του δικαστικού συστήματος ε, των σωμάτων που είναι απαραίτητα για ένα κράτος δικαίου. Θα ήθελα όμως να σας επιστήσω την προσοχή στο εξής. Αυτά που συνέβησαν στο κοσυφοπαίδιο και η επιτυχία του κοσφοπέδιου θα αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες χώρες. Θα αποτελέσει ένα παράδειγμα για τις φιλοδοξίες τις ευρωπαϊκές και θα αποτελέσει παράδειγμα για όλα τα βαλκανικά κράτη. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Μουνής Δεορκίστα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Μία επικοδομητική στάση διαφοροποιημένη όσον αφορά την ανεξαρτησία του κωσιβο πεδίου είχε θετικές αντιδράσεις, γι' αυτό και καταφέραμε να φτάσουμε στη σημερινή πρόοδο. Η Ευρώπη έχει υποφεληθεί και υποφελήθηκε και ολόκληρη η περιοχή από τη σταθερότητα. Αν όλοι είχαμε συμφωνήσει, θα είχαμε πετύχει ακόμα περισσότερα. Ήδη όμως έχουμε πετύχει διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ όλων των πλευρών. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι δεν είναι σωστό η έκκληση που αναφέρεται στην έκθεση ώστε τα κράτη-μέλη που δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσυφοπαίδιο να το αναγνωρίσουν. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι σωστά ούτε όλα αυτά που τα υπόλοιπα που αναφέρονται, τα οποία ε, άρρητα κάπως αναφέρονται. Νομίζω ότι τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το κοσφοπέδιο, η διαφθορά, το οργανωμένο έγκριμα, η οικονομική κατάσταση, η θεσμική οικοδόμηση είναι αυτά που θα πρέπει να υπερτερήσουν και όχι στη συζήτηση και όχι το ποιο έχει αναγνωρίσει το κοσφοπέδιο και ποιο όχι. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Κούκαν τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χάρη, μάλλον ευχαριστώ τον εισηγητή για την ε, έκθεσή του. Θέλω να σας πω ότι υποστηρίζω πλήρως την ατζέντα που έχει ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για φέτος. Η έκθεση σκοπιμότητας, ο διάλογος για την ε, ελευθέρωση των θεωρήσεων είναι πολύ φιλόδοξα βήματα. Βήματα τα οποία επιγόντως ε, χρειάζονται στο κοσυφοπαίδιο σήμερα, όπως λέει και η συγκήτρια. Πρέπει να μπορέσουμε να είμαστε αξιόπιστοι. Θέλουμε αυτά αποτελέσματα και από τις αρχές του κοσυφοπεδίου, ιδιαίτερα στο δικαστικό τομέα, την δημόσια δίκηση, αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε ενίσχυση του κράτους δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά. Θέλω να ενθαρρύνω το κοσυφοπεδίο λοιπόν να συνεχίσει το διάλογο με τη Σερβία προκειμένου να υπάρξουν αυτά αποτελέσματα για τους Κωσοβάρους και προκειμένου επίσης να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Πιστεύω επίσης ότι οι εκπρόσωποι στη συνέλευση του Χρυσοφοπεδίου όμως, και, όπως και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, πρέπει να ενημερωνόμαστε για τη διαδικασία αυτή και για τα αποτελέσματά της. Τέλος, το Κωσυφοπέδιο ε, μένει να κάνει πολλή δουλειά, αλλά έχω εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρει και θα έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά θα ενταχθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα για ένα λεπτό η κυρία Φαγιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την υποστήριξη ενός κράτους που είναι πολύ απομονωμένο στην περιφέρεια αυτή. Ο κόσμος στο κοσφοπέδιο δεν βλέπει ακόμα το φως στην άκρη του τούνελ και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους νέους του Κωσυφοπέδη. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το καθεστώς απελευθέρωσης ε, των θεωρήσεων. Θα πρέπει να δράσουμε γρήγορα και ο διάλογος με τη Σερβία θα πρέπει να σημειώσει ένα βήμα προς τα εμπρός. Μόνο η πλήρης αναγνώριση του 25ου θα επαναφέρει στις φυσιολογικούς ρυθμούς της ζωής Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προετοιμάσει μια τέτοια μελέτη σκοπιμότητας. Οι νέοι χρειάζονται μια προοπτική και θα πρέπει να φροντίσουμε να καταπολεμηθούν το οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά. Όχι μόνο στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά παντού. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί όμω. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Και τελευταίο ο, ο κύριο Φλέκενστάιν. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι ο διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα αποτελεί μια πρώτη επιτυχία εδώ στι Βρυξέλλε. και γι' αυτό ότι αυτό χρειάστηκε θάρρος και τόλμη. Τόλμη του Πρωθυπουργού Τάντιτς και του Προέδρου Τάντιτς. Και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε γιατί αποτελεί ένα πρώτο βήμα, ένα, μια προϋπόθεση για μια θετική εξέλιξη. Τώρα το μπαλάκι είναι σε εμά. Θα πρέπει να δείξουμε στου κοσυφοπέδι ότι έχουμε σοβαρές προθέσεις και γι' αυτό υποστηρίζουμε την Επίτροπο Μάλμστρομ για την δέσμευσή της για την απελευθέρωση από το καθεστώς των θεωρήσεων και γι' αυτό υποστηρίζουμε και τον Επίτροπο Φίλε σε ό,τι αφορά τη μελέτη σκοπιμότητας της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης Θεωροποίηση. Μπορείτε να υπολογίζετε στην αλληλεγγύη μας στο έργο σας αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι στο παρελθόν και στο μέλλον θα πρέπει αμφότερες οι πλευρές να γνωρίζουν ότι μόνο από κοινού και παράλληλα μπορούν να κινηθούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν μπορεί να το πράξει αυτό προς, αν θέλετε, εις βάρος του άλλου. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Έχει το λόγο κύριο Σέρτζο Σιλβέστρης ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λούνατσεκ ε, να τη συγχαρώ για τη δουλειά που μας παρουσίασε. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις και πολλές ευκαιρίες. Ε, εγώ πιστεύω ότι αυτά που πρότεινε σήμερα το Συμβούλιο θα πρέπει να τα στηρίξουμε. Ε, βεβαίως υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία λόγω της προσπάθειας και της πρόοδου που έχει σημειώσει το 25 τα τελευταία χρόνια. Αρκεί να σκεφτούμε ποια ήταν η κατάσταση πριν από 10-15 χρόνια για να καταλάβουμε πόσο σημαντικά βήματα προς τα εμπρός έχουν ήδη γίνει. Σήμερα λοιπόν πρέπει να ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση στην Πρίστινα αλλά και όλες τις πολιτικές πολιτικέ δημοκρατικές δυνάμεις να ακολουθήσουν τον δρόμο της ε, μεταρρύθμισης, ε, να ε, μεταρρυθμίσει τι θεωρήσει στο εμπόριο, στη δικαστική εξουσία και ε, μας περιμένουν δύο στόχοι. Πρώτον, να βελτιωθεί το επίπεδο της δημοκρατίας στο Κοσμοπέδιο, να πλησιάσει το Κοσμοπέδιο στην Ευρώπη και να μπορέσει το Κοσμοπέδιο να ενταχθεί στην Ευρώπη. Πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν μια νέα δημοκρατία η οποία είναι πεπισμένη για τα φιλοευρωπαϊκά της ε, αισθήματα. Πρόεδρος, ε, ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ραμόν Τραβεζές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Το Καταλανικό Κόμμα, από το οποίο προέρχομαι, στηρίζει απόλυτα την προσχώρηση του Κωσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ενώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάμε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν πέντε ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει το Κωσυφοπέδιο σαν μια νέα ανεξάρτητη χώρα. Μία από τις χώρες αυτής είναι η Ισπανία. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συνεχίσουν να πιέζουν την Ισπανία προκειμένου να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του κοσφοπεδίου Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεχτεί αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα μέσα στις ε, χώρες της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κοσφοπέδιο κάνει βήματα προς την ευρωπαϊκή ένταξη μετά από την ανεξαρτησία που διακήρυξε το 2006. Πάντα πρέπει να σεβόμαστε τη δημοκρατία και την ελευθερία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ίνες Κριστίνα Ζούπερ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάντα το λέγαμε και το έχει δείξει και η πραγματικότητα η μονομερής δήλωση ανεξαρτησίας του κοσμοπεδίου είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ σοβαρό προηγούμενο για τη διεθνή κοινότητα και ελοχεύει κινδύνους στην περιοχή και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια παραβίαση της διακήρυξης του Ελσίνκη και ε, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και παραβίαση των αρχών διεθνούς δικαίου. Η δήλωση ανεξαρτησίας ενό ενός ψευδοκράτους δεν ε, είναι κάτι που οδηγεί την περιοχή σε ανεξαρτησία. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια κατοχή. Κάτι το οποίο συμβαίνει με το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ΚΦΟΡ και της ΕΟΛΙΚΣ. Είναι κάτι το οποίο έχει προχωρήσει και σε οικονομική και σε δημοσιονομική κατοχή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Κύριε Ζούμπερ, ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εκτιμώ τις ε, προσπάθειες και τις ε, προοπτικές που ανοίχθηκαν ε, και τις δεσμεύσεις που έχουν δοθεί στον, ε, στην κυβέρνηση του Χάσιν της, αλλά μου φαίνεται ότι ε, δεν σεβόμαστε τις αρχές της ε, ισότητας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης υποδεικνύει τα εγκλήματα της ομάδας Γκρένιτσα στο Κωσίφο Παϊδίο. Εκφοβισμοί, φόνοι των μαρτύρων των εγκλημάτων αυτό, όλα αυτά καταδεικνύουν ότι δεν εκπληρώνονται το έργο δικαιοσύνη στην, ε, στο κοσφοπέδιο και ότι δεν είσαι σε θέση θεωρώ ότι όλες οι ε, κατηγορίες του Συμβουλίου της Ευρώπης θα πρέπει να διερευνηθούν και μόνο τότε θα μπορούσαν να ξανακινήσουν διαπραγματεύσεις με το καθεστώς ε, το οποίο κατηγορείται για βασικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Αγκουστίν Τεμέιρα τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δείχνω την αλληλεγγύη μου στο κοσυφοπέδιο και όταν με επί Μιλόσεβιτς πήγανε στρατόπεδα συγκέντρωσης, στην ίδια μου την πόλη ήρθαν διάφοροι από το Ουτσεκά. Σήμερα όμως, Πρόεδρε, υπάρχουν προβλήματα διαφθοράς στο κοσυφοπέδιο. Έλεγχος των μέσων ενημέρωσης, ε, οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, Πρόεδρε, σήμερα το κοσυφοπαίδιο δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις που πρέπει ούτε για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε για να είναι ανεξάρτητο χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τζαμπασογκάρ, Παρακαλώ. Ε... Míg a 90-es években a koszovói albánok autonómia Ήδη στη δεκαετία του 90 είχαμε μια τελείως διαφορετική κατάσταση στο Κωσφοπαίδιο Και τώρα το Κωσφοπαίδιο έχει γίνει πλέον ανεξάρτητο κράτος. Βεβαίως υπήρξαν πάρα πολλά θύματα και λόγω του πολέμου που έλαβε χώρα. Ε, τα στελέχη της Σερβίας ε, υφάρπαξαν την αυτονομία του Κωσοπεδίου η διεθνής κοινότητα δεν έλαβε σοβαρά υπόψη σε αυτό το σχέδιο του Ρούγκοβα. Ε, θα έπρεπε να γίνει κάτι για να προληφθεί η βία. Βεβαίως ε, υπάρχουν διάφορες εθνοτικές ομάδες σε αυτή την περιοχή και είναι δύσκολο να συνεπάρξουν όλες ειρηνικά. Όμως ε, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να υπάρχει κοινωνική ειρήνη. Δεν ε, νομίζω ότι είναι σωστό να παραπέμπουμε συνεχώς ε, στο παρελθόν ε, σε αυτά που έλεγαν χώρα. Πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι μειονότητες. Πρόεδρος, Ευχαριστούμε για τη διαδικασία Κατσουδιάη. Επόμενη ομιλήτρια. Η κυρία Μπιλμπάου Μπαρανκόντα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις 22 του Ιουλίου του 2010 το Διεθνές Δικαστήριο λέει ότι δήλωση ανεξαρτησίας δεν παραβίασε το διεθνές δίκαιο. Το Κωσεβοπέδιο ήταν χώρα πριν κατακτήσουν το 1912 την περιοχή οι σερβικές δυνάμεις. Και τελικά η υπέστη και τη γενοκτονία του Μιλόσεβιτς. Πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη στα θύματα του σερβικού απεικιοκρατισμού και γι' αυτό πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και έθνη τα οποία θέλουν ένα διαφορετικό καθεστώς. Η Ισπανία πρέπει να καταλάβει ότι τον 21ο αιώνα η βούληση των πολιτών, άπαξ και εκφράζεται ελεύθερα, αποτελεί και τη βάση της κυριαρχίας. Οπότε κύριε Επίτροπε, ποια είναι η γνώμη σα τώρα μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται για να... Ποια είναι η γνώμη σα τώρα για την ένταξη του Κωσυφοπεδίου. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να ζητήσω από τον Επίτροπο Φίλε να πάρει το λόγο. Mr. President, uh, honorable. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, Επίτροπε, ε, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία αυτή για ανταλλαγή απόψεων μαζί σας σε ό,τι αφορά την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κοσυφοπαίδιο. Επίσης, Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξή σα για τι πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προσεγγίσει το 25 την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι αφορά τη μελέτη σκοπιμότητα, ειδικότερα. στου επόμενου μήνε. θα προετοιμάσουμε μια συμβάθο ανάλυση τη της του Κωσυφοπεδίου να συνάψει συμφωνία σταθεροποίηση και σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή θα επιβεβαιώσει την συμμετοχή του Κωσυφοπεδίου μαζί με τα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια, προκειμένου κάποια στιγμή να ενταχθεί στη ζώνη ευημερία και ασφάλειά μα. Η επίσκεψή μου στο Κωσυφοπέδιο αυτή την εβδομάδα σημειώνει, σημείωσε την έναρξη μιας καινούργιας φάσης μεταρρυθμίσεων. Περνώντας από τα λόγια στις ε, διαδικασίες, στην ουσία, στο περιεχόμενο. Αυτό είναι ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπιστούν πολλές προκλήσεις τι πολλέ προκλήσει που αντιμετωπίζει ο λαό του Κωσυφοπεδίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει το Κωσυφοπεδίο στην διαδικασία αυτή. Η πρόσφατη συμφωνία του Κωσυφοπεδίου για την συνεργασία με τη Σερβία αντιμετωπίζοντα πολλά προβλήματα θα πρέπει να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δεσμευτεί ακόμα περισσότερο. Ζήτησα τη διαρκή σα υποστήριξη για να μεταδώσω αυτό το μήνυμα και για να ενισχύσω την δέσμευση και την συνεργασία με το Κοινοβούλιο του Κωσυφοπεδίου προκειμένου να προσεγγίσει και το Κοσμοπέδιο αλλά και όλη η περιφερεια την Ευρώπη και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ευημερία στην, ε, Δυτικά Βαλκάνια. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, εξ ονόματος του Συμβουλίου, ο κύριος, ε, ο Υπουργός, κύριος Βάμεν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Ε, ευχαριστώ την κυρία Λούνα Τσέκ για την στράτευσή της για το κοσυφοπαίδιο και για την, αυτά που μας είπε διαδικασία ένταξης του κοσυφοπαιδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει πάρα πολλές υποχρώσεις απέναντι στο κοσυφοπαίδιο και νομίζω ότι είναι σημαντικό η Γιούλεξ ε, να είναι παρούσα. Βεβαίως ε, την κύρια Φτίνη την φέρουν τα στελέχη του Κοσφοπεδίου ε, που αντιμετωπίζει η χώρα πολλές προκλήσεις. Πολλές εξ αυτών αναφέρθηκαν εδώ. Βέβαια μια τόσο νεοσύστατη χώρα πρέπει να βασίζεται σε ορισμένες προϋποθέσεις. Και το Κοσφοπέδιο σημείωσε μεγάλη πρόοδο αλλά ο δρόμος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύσκολος και ακανθώδης. Πρέπει λοιπόν κανείς ε, να προσπαθήσει, σκληρή δουλειά και ε, το γεγονός ότι πρόσφατα η Σερβία απέκτησε την ε, ιδιότητα της υποψήφιας ε, χώρας. Αυτό κατέδειξε ότι οι χώρες που εκπληρώνουν τις ε, υποχρεώσεις τους έχουν πάρα πολλές και καλές προοπτικές. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι αποτελεί ένα κίνητρο για το οικοσφοπέδιο. Η σημερινή συζήτηση αποτελεί την αφορμή για να εξετάσουμε το μέλλον της χώρας ε, πρέπει να πούμε ότι η πρόοδο ε, σε ορισμένου τομεί, κυρίω ε, στη διαφθορά και στην αντιμετώπιση του εγκλήματο, είναι περιορισμένη. Αυτή η διαφθορά είναι πραγματικά πρόβλημα. Θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη πρόοδο. Και όταν εξαιρούνται μάλιστα ορισμένα θέματα όσον αφορά τα ποινικά κολάσιμα δικήματα, ούτε αυτό είναι καλό. Όσον αφορά επίσης ε, την, ε, το οργανωμένο έγκλημα, πρέπει να θεσμιστούν ε, νομοσχέδια και να εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες πρέπει να λαμβάνει χώρα γιατί το έγκλημα είναι διασυνοριακό. Ε, σε τελική ανάλυση το νομικό και δικαστικό σύστημα πρέπει να μεταρρυθμιστεί στο κοσμοπέδιο και εκεί θα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την οικονομία χρειαζόμαστε ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, που θα μετατρέψουν το κοσμοπέδιο σε ε, οικονομία της αγοράς, οι προκλήσεις είναι μεγάλες, ε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούται να βοηθήσει, όπως σας είπα, αυτό το νεοσύστατο κράτος έτσι ώστε και αυτό να μπορέσει να πλησιάσει περισσότερο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Κωσοβάροι επιθυμούν να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το διάλογο διαπίστωσε ότι ακόμα και αν είναι δύσκολη η περιραίους ατμόσφαιρα μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος. Ελπίζω λοιπόν η ε, κυβέρνηση στην Πρίστινα να προχωρήσει ρεαλιστικά ε, και να συνεχίσει να προσπαθεί να ε, βελτιώσει την κατάσταση στο Κοσμοπέδιο. Η Ιδανική Προεδρία θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Ε, θέλω να σας πω ότι πήρα μία πρόταση ψηφίσματος, ε, έληξε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 11.30.